θέτημα για την απαγόρευση της ομοφιλοφιλίας. Για πρώτα ο κύριος Κάσμαν από πλευράς των συντακτών θα λάβει τον λόγο. Κύριε Κάσμαν, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ζητώ την ε, ε κατανόηση της ε, συνέλευσης εδώ να φύγουμε από το διαδικαστικά και να πάμε ε, στο θέμα αυτό της διακριτικής μεταχείρισης. Κάποιος ε, μπορεί να πει τι μας αφορά μια νομοθεσία του Κοινοβουλίου της Ουγκάνας. Αλλά κάθε παραβίαση ανθρώπινου δικαιώματος έχει σχέση και μας αφορά. οποιοδήποτε άτομο, λέει ο νόμος αυτός που υποτίθεται ότι είναι ομοφιλόφιλος, κινδυνεύει να καταδικαστεί σε ισόβια φυλάκιση. Ε, Όποιος δεν καταγγέλει ε, λεσβείε ή ομοφυλόφιλους ε, απειλείται με ε, φυλάκιση ή πρόστιμα. Πρέπει ο καθένας να καταγγέλει ε, οποιονδήποτε ομοφυλόφιλο κλπ. μέσα σε 24 ώρες. Ε, ε, σπιτονικοκύρης που νοικιάζει το σπίτι του σε υπο σε ύποπτο για ομοφυλοφιλία και δυνεύει με φυλάκιση 7 ετών. Αυτό μπορεί να καταστρέψει την ε, φήμη οποιοδήποτε που δουλεύει με τέτοιο πληθυσμό, όπως γιατροί, ε, ε, οργανώσεις κοινωνιών των πολιτών, όλους αυτούς που εργάζονται στην, στην τομέα, στον τομέα της αναπαραγωγικής υγείας. Και ο νόμος αυτός θα διευκολύνει την διάδοση του ιού του AIDS. Πρέπει να υπερασπιστούμε αυτού του ανθρώπου που δεν έχουν κανέναν να υπερασπιστεί τα δικαιώματά του. Ο κύριος, ε, ο Τεμπρούκ έχει κάνει σχετική ε, δήλωση. Ε, η γαλλική κυβέρνηση, η σουδική κυβέρνηση, ο πρόεδρος Ομπάμα και οι εκπρόσωποι της, του Υπουργείου Εξωτερικών. Ε, πρέπει να δώσουμε στο θέμα αυτό ε, τη σημασία που του ε, αξίζει ώστε να ακουστεί η φωνή των ανθρώπων στην Ουγγάντα που δεν γίνεται ακουστή σήμερα. Κάσμαν, τώρα πάλι από τους συντάκτες του ψηφίσματος η κυρία Σάκε. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο και τους συναδέλφους που παρίστανται εδώ. Πέρυσι το Σεπτέμβριο ένα, ένας βουλευτής από την Ουγκάντα ε, υπέβαλε ένα ε, νομοθέτημα κατά της ομοφιλοφιλίας που προβλέπει ως κύρωση μέχρι και τη θανατική ποινή. Δεν αναφέρεται μόνο στους ε, υπόπτους ως εγκληματίας αλλά και άτομα τα οποία προσφύζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα ή στην Ουγγάντα. Οπότε κατά αυτόν τον τρόπο παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και ε, διεθνείς παγκόσμιες αξίες. Απορρίπτουμε την ποινή της θανατικής ε, ποινής και επίσης ε, ανησυχούμε πολύ για τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις οι οποίες ενδέχεται να καταργήσουν τις δραστηριότητες τους στην Ουγγάντα και συμφωνούμε με όσους ζητούν να καταδικαστούν αυτό το ε, νομοθετικό σχέδιο και το, νομοσχέδιο και ε, να ε, ενημερωθεί η Ουγγάντα. Ευχαριστώ για ένα λεπτό και πάλι ο κύριος Τάνεκου. Κύριε Πρόεδρε, ε, η Ουγγάντα είναι μία παραδοσιακή χώρα. Η ομοφιλοφιλία είναι παράνομη όπως και σε πολλές χώρες της Αφρικής. Πρέπει να είμαστε ευαίσθητοι όταν θέλουμε να επιβάλλουμε τις πιο ανεκτικές και φιλελεύθερες αξίες μας στους άλλους. Αλλά πρέπει βεβαίως να κατακρίνουμε αυτό το νομοσχέδιο το οποίο είναι δρακόντιο και υπερβολικό όχι μόνο θα είναι εις βάρος της ασφάλειας των ομοφιλοφίλων στην Ουγκάντα αλλά θα αμαυρώσει την εικόνα της Ουγκάντας διεθνώς και θα την καταστήσει παρία. Τις δύο τελευταίες δεκαετίες έχει διαμορφωθεί σε ένα πρότυπο ε, της ε, αναπτύξεως στην Αφρική Ουγκάντα. Γιατί λοιπόν τώρα ε, πρέπει η χώρα τους να τοποθετηθεί ε, δίπλα στο Ιράν το οποίο καταδικάζει και εκτελεί δημοσίως τους ομοφιλοφίλους. Μία τέτοια άγρια νομοθεσία ε, δεν μπορεί να προχωρήσει και θα πρέπει να ζητήσουμε από την Ουγγάντα να το απαγορεύσει. Ευχαριστώ και ε, η επόμενη είναι η κυρία Λούνατσεκ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήδη από τους προλαλήσαντες ήδη έχουν ε, διαγράψει τις λεπτομέρειες του νομοσχεδίου που υπάρχει στην Ουγκάντα. Θα ήθελα να σας, να σας διηγηθώ μία ε, ιστορία. Ήμουνα πριν 4-5 ε, χρόνια εις τη Καμπάλα και συνάντησα ομοφιλόφιλους άντρες και γυναίκες εις την, σε μια πιτσαρία της Καμπάλα. Και έχθη στη συνέχεια ότι πρόκειται να υπάρξουν διωγμοί ε, στις περιοχές όπου συχνάζουν οι ομοφυλόφιλοι ε, και εγώ φοβόμουν εκείνο το βράδυ δεν συνέβη τίποτα αλλά έχει ξεκινήσει μία ε, ομοφιλοφοβία στην Ουγγάντα όπου τιμωρείται όχι απλώς το γεγονός αυτό αλλά διατάσσεται και ανθρώπινη και ποινή ε, ε, καταδείξη θάνατον. Υπάρχουν τέτοια προβλήματα σε πολλές χώρες. Να λέμε τώρα όμως ότι η ομοφιλοφιλία δεν είναι αφρικανική είναι λανθασμένο. Ε, δεν, πρόκειται για ένα γεγονός που υπάρχει ασχέτως νομοθεσιών και χαίρομαι διότι όλες οι πολιτικές ομάδες έχουν καταρτήσει ένα κοινό ψήφισμα πράγμα το οποίο θα επιτρέψει να ενισχύσουμε όλους τους ομοφιλόφιλους στην Ουγγάντα και να μην τους καταδικάζουμε. Σαν Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ε, την υποχρέωση να διακηρύσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα παντού και να τονίσουμε ότι στη Συμφωνία του Κοτονού ο, περιλαμβάνονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και η προάσπισή τους για όλους και παντού. Ελπίζω ότι το ψήφισμα όπως έχει παρατεθεί θα μπορέσει να υιοθετηθεί διότι οργανώσεις οι οποίες είναι υπέρ των ε, δικαιωμάτων των ομοφιλοφίλων θα πρέπει να συλληφθούν επίσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από όλους τους άλλους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε συνάδελφε Λούνατσεκ. Και ως συντάκτεια τώρα η συνάδελφος Στίφρε παρακαλώ. Ναι κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Το θέμα που απασχολεί το Ευρωκοινοβούλιο είναι η νομοθεσία αυτή στην Ουγγάντα που παραβιάζει τα θεμελιώδη ανθρώπινη δικαιώματα και δεν πρέπει για κανένα τρόπο να ε, εγκριθεί. Η ε, ποινικοποίηση της ομοφιλοφιλίας ε, αν εγκριθεί αυτός ο νόμος το 2010 θα επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο η κατάσταση και θα μπορεί η ομοφιλοφιλία να καταδικάζεται ε, με ισόβια φυλάκιση ή και με θανατική ποινή για τους οροθετικούς ε, Αυτό είναι ό,τι καλύτερο για την περαιτέρω διάδοση του AIDS. Ε, όπως είπε ο κύριος Κάσμαν, εξάλλου ο νόμος υποχρεώνει τους πολίτες να καταγγείλουν μέσα 24 ώρες ένα ομοφιλόφιλο. Αν είναι κανείς δάσκαλος, γιατρός, γόνιος, πρέπει να καταγγείλει την ομοφιλοφιλία ε, ποινή φυλάκισης. Ε, επίσης, ε, αυτό ε, αφορά τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, όλους τους, ε, όλες τις οργανώσεις των πολιτών που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ουγγάντα. Διακόπτει ο Πρόεδρος. Αγαπητή συνάδελφος, όταν, αν μπορώ να σας παρακαλέσω να μην τρέχετε τόσο πολύ, μιλάτε πιο αργά παρακαλώ. Μόλι υποβλήθηκε το νομοσχέδιο αυτό στο Κοινοβούλιο της Καμπάλα, καταδικάστηκε ε, ταυτόχρονα από ολόκληρο τον κόσμο, η Γαλλία, οι Ηνωμένε Πολιτείε, ο Ευρωπαίος ε, Επίτροπος κ. Τεκιού, καταδίκασαν το νέο αυτό νομοσχέδιο. Η Ουγγάντα πρέπει να σεβαστεί τι διεθνεί υποχρεώσει τη και τη Συμφωνία του Κοτονού. Είναι επίγον η Ευρωπαϊκή Ένωση να προβεί σε διαβήματα ενώπιον των αρχών τη Ουγγάντα και να ε, ξανασκεφτεί τι σχέσει τη και τι δεσμεύσει απέναντι στη χώρα αυτή, αν συνεχιστεί και προωθηθεί αυτό το νομοσχέδιο. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφε, 12 δευτερόλεπτα θα είχατε ακόμα χρόνο αν διαβάζατε με αργότερο βραδύτερο ρυθμό, τότε οι περισσότεροι συνάδελφοι θα υποφελούν από καλύτερη διερμηνία. Για όσους διαβάζουν, θα πρότεινα να διαθέτουν, όσους έχουν έτοιμο κείμενο, να το διαθέτουν στους διερμηνείς. Βοηθά αυτό στην ποιότητα διερμηνίας. Επόμενος από τους αγορητές συντάκτες, Κάτσμαρεκ, ένα λεπτό για το ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κάτι με το οποίο δεν θα έπρεπε να ασχοληθούμε είναι το θέμα αυτό, διότι η περάσπιση των δικαιωμάτων των ομοφιλοφίλων δεν δικαιολογείται. Είναι μια επέκταση και διεύρυνση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όμως αυτό δεν αληθεύει διότι τα δικαιώματα όλων μπορούν να επικαλούνται εδώ και κανένα δεν μπορεί να αποκλείεται. Δεν είναι νέο θέμα ο σεξουαλικός προσανατολισμός και οι σεξουαλικές επιλογές. Θα πρέπει όμως να συμφωνηθεί ότι τέτοιου είδους παραβιάσεις είναι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για εκείνου που ενδιαφέρονται για αυτό το θέμα και εμπλέκονται με αυτόν τον τρόπο λένε πολλοί ότι έχουμε ένα νέο νέο ε, απεικιοκρατικό τρόπο σκέψης και επιβάλλουμε τις απόψεις μας στους άλλους. Ούτε και αυτό αληθεύει όμως. Δεν ε, γίνεται αυτό από εμά. Εκτιμούμε και σεβόμαστε την ανεξαρτησία τη ε, Ουγγάντα και τα κυριαρχικά τη δικαιώματα. Δεν πρέπει να αγνοούμε μια τέτοια κατάσταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, συνάδελφε Κάσμαρεκ. Συνέχεια ο κύριο Σαρίφ, εξ ονόματο τη ΕΣΔΕ, παρακαλώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, χαίρομαι που αναφέρεστε ή σε το νομοσχέδιο που ε, ε, υπευλήθη ή στο Κοινοβούλιο της Ουγγάντα το Σεπτέμβριο διότι νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πέραν του ότι χωρίζει τις πολιτικές οικογένειες να ζητήσει να καταδικαστεί αυτό το σχέδιο και να αναθεωρηθεί η νομοθεσία που ποινικοποιεί την ομοφιλοφιλία Όπω Όπως είπε ο κύριος Κάσμαν και οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις έχουν καταφερθεί κατά αυτού του νομοσχεδίου. Ο Επίτροπος και πολλά κράτη καθώς άλλωστε και οι δηλώσεις του Προέδρου Ομπάμα καταδικάζουν αυτή την πρωτοβουλία. Θα έλεγα λοιπόν ότι πρέπει να, εάν δεν ανακληθεί, να αναθεωρήσουμε τις δεσμεύσεις μας προς την Οργάντα διότι δεν μπορεί κανείς να συνεχίσει να χαίρει της βοηθείες Ευρωπαϊκής Ενώσεως εάν καταπατά τα, τις συμφωνίες του Κοτονού. Και επίσης κανείς δεν πρέπει να κροτηριάζεται ή να βασανίζεται και δεν μπορεί να υπάρξει θέμα από αυτού. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και τώρα για την ομάδα των Προέδρων για τρία λεπτά ο κύριος Μέντα Ερουέντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε δεν ε, μπορούμε να συζητήσουμε για την ε, ε, περίπτωση της αμήνα του Χαϊντάρ για λόγους που όλοι ξέρουμε. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα αυτό της Ουγκάντα έχει τραβήξει την προσοχή μας και συζητάμε ακόμη μια φορά το θέμα της ομοφοβίας. Στο παρελθόν έχουμε υιοθετήσει διάφορα ψηφίσματα για τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Σήμερα προστίθεται ένα ακόμα τέτοιο ψήφισμα. Ε, χρειάζεται μια πολιτική απάντηση στο νομοσχέδιο αυτό της Ουγκάντα. Ε, η διακριτική ε, μεταχείριση εις βάρος αυτών που υποτίθεται ότι είναι λεσβείε, ομοφιλόφιλοι, ομοφιλόφιλοι πανεδηματίες, που οι ποινές μπορούν να φτάνουν μέχρι και την θανατική ποινή ή μέχρι και τρία χρόνια φυλάκιση για όποιον παραλείπει να καταγγείλει οποιοδήποτε γνωρίζει ότι ανήκει σε αυτές τις ομάδες. Αυτό σημαίνει ότι οποιοδήποτε, ο καθένας από εμά θα μπορούσε ε, να ε, συρθεί στη φυλακή για κάποιον από αυτούς τους λόγους. Πρέπει να υπενθυμίσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους διεθνείς οργανισμούς ότι το, η ελευθερία του γενετήσιου προσανατολισμού διέπεται από το διεθνές δίκαιο και βάσει αυτού πρέπει να μην υπάρχει διακριτική μεταχείριση και να εξασφαλίζεται η ελευθερία επιλογής. Οι διεθνείς δωρητές, κυβερνητικοί και εμεί πρέπει να σταματήσουν τις δραστηριότητές τους στη χώρα αυτή αν περάσει αυτό το νομοσχέδιο και ε, βεβαίω πρέπει να είμαστε ριζικά αντίθετοι σε κάθε απόπειρα εισαγωγή τη θανατική ποινή. Αν δεν συμμορφωθούν οι αρχέ τη Ουγγάντα, πρέπει το Συμβούλιο και η Κομισιόν να ξανασκεφτούν τι σχέσει του και τι δεσμεύσει με την ε, Ουγγάντα όταν η χώρα αυτή ε, παραβιάζει τι ε, υποχρεώσει όσον αφορά το διεθνέ δίκαιο. Πρέπει να υπενθυμίσουμε στην κυβέρνηση τη Ουγγάντα τι διεθνεί τη υποχρεώσει και τη συμφωνία του Κοτονού. Τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να γίνουν σεβαστά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ρομέντε Ρουέντα. Τώρα η κυρία Γκόμες για ένα λεπτό. Η Ευρώπη πρέπει να παρέμβει σε αυτό το θέμα όσον αφορά την συμφωνία, το πλαίσιο συμφωνής Κοτονού πρέπει να ζητήσουμε άμεσα την κατάργηση αυτού του νομοθετήματος. Διαφορετικά θα υπάρξουν επιπτώσεις στην ε, πολιτική ε, συνεργασία με την ε, Ουγγάντα. Όταν είδαμε και βλέπουμε την θλιβερή μοίρα των ομοφιλοφίλων στην Ουγγάντα και στο Ιράν και σε άλλες χώρες βλέπουμε πόσο βλέπουμε ότι σε πολλούς πολιτισμούς υπάρχει ένα, μια παραβίαση δεσμεύσεων και υποχρεώσεων όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και εδώ βλέπουμε και τον ρόλο της ε, ακροδεξιάς ε, των Ευαγγελιστών Αμερικανών ε, αναλαμβάνοντας τέτοιου είδους δραστηριότητες στην Αφρική. Η Ευρώπη, όλη, η Ευρώπη πρέπει να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της επιτόπου στις χώρες αυτές για να καταπολεμήσει το σκοταδισμό και την τάση αυτή να επιβάλλονται, ας το πω έτσι, ως εγκλήματα οι επιλογές της, του σεξουαλικού προσανατολισμού. Ευχαριστώ. Στη συνέχεια Γιάννης Μπαριονουέβο ε, Γκαρσία παρακαλώ, ένα λεπτό. Εκφράζω την ικανοποίησή μου, Πρόεδρε, για την ομοφωνία που εκφράζουν οι συνάδελφοι διαφορετικών ομάδων για αυτό το Ουγγαντέζικο νομοθέτημα το οποίο προκαλεί και καταδικάζεται από εμάς ομόφωνα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το μόνο αίτημα για να ζητήσω τον λόγο είναι να εκφράσω εγώ διαζώσεις ε, με τη φωνή μου αυτή την άποψη και μετά θα ψηφίσω. Προσθέτω τη φωνή μου στον Μάικλ Κάσμαν, στη φωνή του Μάικλ Κάσμαν και στους εκπροσώπους της ομάδας ε, διότι ο αγώνας ε, κατά της μυσαλλοδοξίας και κατά της ε, και κατά της θανατικής ποινής ε, πρέπει να μας κάνει να είμαστε πολύ στεναροί και να ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο και εκείνη να είναι στεναροί απέναντι στην ε, Ουγγάντα ώστε να καταργηθεί αυτό το νομοθέτημα και έτσι να καταφέρουμε η Ουγγάντα να μπορέσει να επανορθώσει. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Μπαριονούεβο Γκαρτία. Περνάμε τώρα στη διαδικασία Catch the Eye. Πρέντας έχει τον λόγο, παρακαλώ, συνάδελφος. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να σας πω ότι ε, είμαι πάρα πολύ ενοχλημένος από αυτή την απαράδεκτη νομοθεσία η οποία ε, ποινικοποιεί την ομοφιλοφιλία και την, ε, ε, ε, και τη συγκάλυψη πληροφοριών για τη σεξουαλική δραστηριότητα των ατόμων. Ιδίω διότι εδώ μιλάμε για μία δεύτερη αναθεώρηση της συμφορίας του Κοτονού την οποία έχει προσυπογράψει και η Ουγγάντα. Η συμφωνία αυτή προβλέπει την ε, ανάγκη ε, σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτή την εβδομάδα ε, έγινε μία έκθεση από την κυρία Ζολή σχετικά με την συνθήκη του Κοτονού. Και ήδη χάρη σε αυτό το έγγραφο ξέρουμε ποια είναι τα συμφραζόμενα για κάτι το οποίο καταδικάζουμε. Ευχαριστώ η κυρία Πρέντα τελευταία και μετά η κυρία Ρουτέλα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να προσθέσω το εξής του χρόνου το Μάιο ή στην Καμπάλα, στην Ουγγάντα, θα γίνει ένα συνέδριο το οποίο θα, θα αναθεωρήσει την ε, θέση των ΡΟΜ ε, για να μπορέσει ε, να ανανεωθεί η θέση στο, στο Διεθνές Δικαστήριο και εκεί θα πρέπει να ξανασυζητηθεί και όλη ε, η, η, σχετική νομοθεσία. Ευχαριστώ τώρα ο Επίτροπος κύριος Ζαμέτσκι. Ε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η Επιτροπή ανησυχεί πάρα πολύ για αυτό το νομοσχέδιο το οποίο υπευλήθη το Κοινοβούλιο της Ουγάντα και επεμβαίνει σε βασικά θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ανησυχούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία θεωρεί ότι η ποινικοποίηση της ομοφιλοφιλίας που προβλέπεται εις ε, το νομοσχέδιο παραβιάζει την ε, ε, συνθήκη για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην οποία έχει προσυπογράψει η Ουγγάντα. Θα πρέπει λοιπόν να ακολουθήσει και να συμμορφωθεί με τις διεθνείς της υποχρεώτης η Ουγγάντα ακόμη και στο θέμα των, ανθρωπι... των ε, σεξουαλικών δικαιωμάτων και να απογονικοποιήσει την ε, ε, ομοφιλοφιλία. Το θέμα αυτό είχε παρουσιαστεί στον κύριο Μουσελένη πέρυσι τον Νοέμβριο διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποδίδουν μεγάλη σημασία κύριος αυτός είχε, είχε εκφράσει την πεποίθησή του ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει μία τέτοια νομοθεσία. Ο πρόεδρος έχει θέσει το θέμα με ε, τον, ε, με τον Υπουργό Δικαιοσύνης της Ουγγάντα και την κυβέρνηση. Στο τελευταίο διάβημα την 3η ε, Δεκεμβρίου ο υπεύθυνο των εξωτερικών σχέσεων επιβεβαίωσε την στήριξή του στις θεμελιώδεις ελευθερίες και θύμισε στην Ουγγάντα ε, τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει. Ο υπουργό ε, ε, απάντησε ότι χρειάζεται χρόνος για να αλλάξουν οι συνθήκες και υπάρχουν άτομα τα οποία προσιλητίζουν τους νέους σε ομοφιλοφιλία. Ε, ζήτησε λοιπόν να παρακολουθήσει ο ίδιος ε, μέσω του Υπουργικού Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου το θέμα για να μπορεί να επέμβει σωστά. Ε, η συνεργασία με την Ουγγάντα κατά τη γνώμη της Επιτροπής ε, θα οδηγήσει σε ε, μία αναθεώρηση της σχετικής νομοθεσίας η οποία θα πρέπει να συνάδει με την αρχή της κατάργησης των διακρίσεων ασχέτως των σεξουαλικών προσανατολισμών. Ευχαριστώ κύριε Ζαμίνσκι. Έληξε η συζήτηση του θέματος αυτού και στο τέλος των συζητήσεων θα γίνει ψηφοφορία. Τώρα έχουμε 7 ε, ψηφίσματα για το Αζερβαϊτζάν σχετικά με την ελευθερία της ε, έκφρασης και πρώτος ο κύριο Προβέρα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ